από κοινού, από το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν, ε, καθώς θα εκτιλήσετε η στρατηγική μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνω τη συζήτηση. Θα ψηφίσουμε επί του κειμένου την Δετάρτη στις 12.30. Ξεκινούμε τώρα τη συζήτηση για την έκθεση Κόχ και Σενάλεβα για την ηλεκτρονική κλίση, μια νέα υπηρεσία 112 για τους πολίτες. Να δώσω το λόγο στους δύο εισηγητές, τέσσερα λεπτά στον καθένα. Ο κύριος Δίτερ Κόχ, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, χιλιάδες άνθρωποι θα μπορούσαν να είναι ακόμα στη ζωή ή δεν θα είχαν μόνιμες αναπηρίες αν μετά το ατύχημα γρήγορα ε, μέσα στην πρώτη χρυσή ώρα όπως το λέμε θα μπορούσαν να είχαν τύχει ε, επαγγελματικής ιατρικής βοήθειας. Τώρα το όραμα αυτό το προσεγγίζουμε περισσότερο. Ε, το οίκολ που συζητάμε δεν μπορεί να προλάβει τα αρχαία ούτε αποσυνδέει από, τις πρώτες, από την ανάγκη για πρώτες βοήθειες, βοήθειες. Όμως αυτομάτως ενημερώνει σημαντικές αρχές. Ε, προφανώς ε, θα πρέπει να αποφύγουμε ε, καταχρήσεις, υπερβολική χρήση. Αυτό θα γίνει μαζί με τους κατασκευαστές. Ε, υπάρχουν γιατροί ε, πρώτων βοηθειών που μπορούν να αποστέλλονται μετά από το, το αυτόματο τηλεφώνημα. Η υλοποίηση θα πρέπει να γίνει από τα κράτη-μέλη το, σύστημα e-call ε, μέχρι ε, όταν δεν ε, υπάρχει τροχαίο είναι ενυπνώση θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι πολύ καλύτερο από ένα κινητό διότι είναι αυτοματοποιημένο. Ε, μπορεί επίσης ε, να ενεργοποιηθεί ε, και χειρονακτικά και στέλνει πολύ σημαντικές πληροφορίες σε ομάδες διάσωσης. Έτσι, επίσης τα δεδομένα αυτά αναγνωρίζονται ως κατεπήγον τηλεφώνημα και αντιμετωπίζονται έτσι. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει τις υπηρεσίες διάσωσης να τις βελτιώσουν, να τις αναβαθμίσουν. Αυτό το σύστημα e-call θέλουμε να χρησιμοποιείται ε, με το, στο 112, το οποίο είναι διεθνής αριθμός, θα χρησιμοποιείται και θα εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη και επίσης είναι και συμβατό με τα συστήματα των τρίτων χωρών. Ε, είναι ένα σύστημα το οποίο στηρίζεται σε ουδέτερη αρχιτεκτονική δεδομένων. Επίσης μπορεί αργότερα να συνδεθεί και με ε, άλλα συστήματα όπως διαθεσιμότητα, θέσεων, πάρκινγκ κλπ. ή και με τις ε, δημόσιες μεταφορές. Αυτό το θα πρέπει να ε, ε, εφαρμόζεται σε ιδιωτικό και σε δημόσιο επίπεδο. Οι χρήστες ε, πάνω στη βάση των διεξοδικών πληροφοριών θα μπορούν να επιλέγουν ένα τέτοιο σύστημα το οποίο μπορεί να είναι παράλληλο ε, και με άλλα συστήματα ασφαλιστικά κλπ. Ε, το 80% των ε, οδηγών επιθυμούν ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο άλλωστε το καλωσορίζουν και το προωθούν και θύματα τροχαίων. Δεν επιτρέπεται λοιπόν να το καθυστερούμε εμείς. Αύριο περιμένω να τύχει έκθεση ευρείας υποστήριξης. Ευχαριστώ. Η κυρία Σενάλοβα. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, Αυτά είναι θέματα που προκαλούν πάρα πολύ ζωηρές συζητήσεις. Πέρασαν χρόνια από τότε που συζητήσαμε το θέμα των ε, ζωνών ασφαλείας Είμαστε στο 2012 και μιλάμε για περαιτέρω στοιχεία που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την παθητική ασφάλεια στου ευρωπαϊκού ε, δρόμου. Πρόκειται για το σύστημα ηλεκλήσης. Τι είναι το e-call. Πρόκειται για ένα σύστημα που σε περίπτωση ατυχήματος καλύπτει με το, το 112 την αρμόδια υπηρεσία. Το e-call ενημερώνει τους διασώστες άμεσα για το σημείο όπου έγινε το ατύχημα και δεν υπάρχουν και γλωσσικά εμπόδια για να γίνει αυτή η κλίση. 2.500 ατυχήματα λιγότερα, το 15%, 15 λιγότερη τραυματίας. Είναι λοιπόν σαφή σαφείς επιχειρήματα. Γιατί όμως ε, αυτά δεν εφαρμόστηκαν. Η εισαγωγή της ε, ηλεκλήσης σε όλες τις χώρες ε, αποτέλεσε μία από τις βασικές προτεραιότητες που έτυχαν αναγνώριση στο 2002 πρακτικά. Διαπιστώθηκε ότι είναι καλύτερα μία θελοντική εφαρμογή του συστήματος. Αυτό δεν είναι ε, ε, αποτελεσματικό. Μόνο αυτοκίνητα ανώτατης κατηγορίας έχουν ένα σύστημα που μπορεί να αντικαταστήσει το σύστημα e-call και να καλύψει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή πέρσι πρότεινε τρία έγγραφα Μέχρι στιγμής όμως έχει δημοσιευθεί μόνο ένα, μία σύσταση του 2011 για τις χώρες μέλη και για τους ε, φορείς κινητής ε, τηλεφωνίας. Το δεύτερο έγγραφο, σύμφωνα με την Επιτρόπο Κρούς, θα έπρεπε ήδη να δημοσιευθεί το πρώτο τρίμηνο αυτού του έτους. Αυτό θα ήταν το πρώτο νομοθετικό βήμα για την υποχρεωτική εφαρμογή του συστήματος e-call. Είμαι πεπισμένη συνεπώς ότι αύριο θα επιβεβαιώσουμε την κοινή θέση των Επιτροπών Τραν και Ίκο και ότι η Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποστηρίξει την υποχρεωτική εφαρμογή του συστήματος Θα εκμεταλλευτούμε τη δυνατότητα να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στην Επιτροπή. Δηλαδή οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εφαρμογή εφαρμογή του e-call δεν είναι πλέον ανεκτή. Οι νομοθετικέ προτάσει θα πρέπει να υποβληθούν το σύντομο των δυνατών έτσι ώστε όλοι οι πολίτε από το 2015 να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτέ τι κλήσει έκτακτη ανάγκη με το 112 του 112 σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το e-call θα πρέπει να είναι δωρεάν για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα οχήματα ανεξάρτητα από την μάρκα ή από την τιμή τους, τη τιμή αγοράς του. Σήμερα Συμπερασματικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κοχ και όλους τους συναδέλφους καθώς και τη γραμματεία και τους βοηθούς μας για τη συνεργασία που οδήγησε στη διατύπωση αυτής ε, της έκθεσης που στέλνει ένα πάρα πολύ σαφές μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Προχωρούμε με τη διαδικασία Catch Πάρα πολλοί έχουν ζητήσει το λόγο. Δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο σε όλους. Να ξεκινήσω με την κυρία Ροϊτόβα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ως γιατρός γνωρίζω ότι σε σοβαρές περιπτώσεις τροχαίου ατυχήματος παίζουν ρόλο ακόμα και τη δευτερόλεπτα. Προσπαθούμε λοιπόν το σύστημα αυτό να το εντάξουμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο ένα ολοκληρωμένο σύστημα μας επιτρέπει να δράσουμε έγκαιρα και άμεσα επιτρέπει να αποφύγουμε τα λησιωτά ατυχήματα. Ορισμένα αυτοκίνητα ήδη επιτρέπουν τη χρήση αυτής της υπηρεσίας. Για παράδειγμα στη Γερμανία. Χαίρομαι ιδιαίτερα που αυτό το σύστημα θα γίνει υποχρεωτικό επιτέλους σε δύο χρόνια. Αυτό το ευρωπαϊκό δωρεάν σύστημα θα είναι το μοναδικό απτό παράδειγμα τη θέμενης αξίας της ολοκλήρωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελπίζω η Επιτροπή να κάνει ό,τι καλύτερο για να υποβάλει τις προτάσεις της. Ευχαριστώ κυρία Ζήτα Γκουρμάη. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, να ευχαριστήσω τους εισηγητές και τους συναδέλφους στην Αρμόδια Επιτροπή για τη συνεργασία τους. Θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα που να σώζει ζωές σε όλα τα νέα αυτοκινήτα από το 2015 και μετά. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει την πρόταση για την ηλεκτρονική κλίση σε λιγότερο από το 1% των ε, ιδιωτικής χρήσης επιβατικών οχημάτων αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ε, το σύστημα αυτό, το οποίο στοιχίζει λιγότερο από 240 ευρώ και μπορεί να σώσει πάνω από 2.500 ζωές και παραπάνω ε, ετησίως. Και γι' αυτό ε, θα πρέπει πάντοτε να στηρίζεται στον αριθμό κλήσης επίγουσας ανάγκης. Να είναι υποχρεωτικός ο χαρακτήρας της εφαρμογής του συστήματος από το 2015 και μετά. Αυτό είναι η πρότασή μας. Είναι κάτι που θα ωφελήσει τους πάντες. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, η κυρία Σινκλέρ. Και αν δεν είναι παρούσα, η κυρία Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα της έκθεσης αυτής είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το νέο σύστημα διευκολύνει τη διάσωση όλο και περισσότερων Ευρωπαίων πολιτών οι οποίοι μπορεί να πάθουν κάποιο ατύχημα. Επομένως, η προστιθέμενη αξία που θα έχει αυτό το σύστημα θα εξαρτηθεί από την υπεύθυνη στάση που θα υιοθετήσουν τα κράτη-μέλη. Και θέλω να σας ενημερώσω για τις δραστηριότητες της Σλοβακίας ως προς αυτό. Έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα για την κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού διάσωσης. Η κατάρτιση είναι σημαντική έτσι ώστε ε, οι διασώστες να λειτουργούν σωστά και το σύστημα να δουλεύει. Οι διασώστες λοιπόν έχουν, κάνουν κατάρτιση στην τεχνολογία της επικοινωνίας και των πληροφοριών και λαμβάνουν κατάρτιση στις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στις περιφερειακές γλώσσες. Στην κατάρτισή τους παρακολουθούν μαθήματα επικοινωνίας και έχουμε αξιοποιήσει και ευρωπαϊκά κονδύλια ε, με το σκοπό αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Φίλε Μπρέντερκαστ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι τα οδικά ατυχήματα ε, επιβάλλουν ένα πολύ μεγάλο φόρο αίματος στις κοινωνίες μας και αυτό το σύστημα πράγματι θα σώσει ζωές. Δυστυχώς ενώ είναι προτεραιότητα τα τελευταία δέκα χρόνια ε, λειτουργεί σε πολύ περιθωριακό βαθμό και είναι μόνο στα αυτοκίνητα υψηλής κατηγορίας προς το παρόν. Ευχαριστώ τους εισηγητές για τη δουλειά τους. Στηρίζω την πρότασή τους ε, να είναι υποχρεωτική και δωρεάν η κλίση στο 112 σε όλα τα αυτοκίνητα από το 2015 και μετά. Θα πρέπει να νομοθετήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση για να έχουμε οικονομίες κλίμακας και οικουμενική υιοθέτηση αυτού του συστήματος. Και είναι κάτι που θα ωφελήσει κυρίως και την ύπεθρο, της αγροτικές περιοχές. Θα μειωθεί ο χρόνος ανταπόκρισης στο μισό ειδικότερα σε τέτοιου είδου περιοχές που είναι πολύ δύσκολο ο ακριβής προσδιορισμός της γεωγραφική θέσης του αυτοκινήτου. Γι' αυτό και εγώ προτείνω η εφαρμογή του συστήματος αυτού να είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Τιτσάο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, θα ήθελα να πω ότι 31.000 άνθρωποι πέθαναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε 1,15 εκατομμύρια οδικά ατυχήματα. Η εισαγωγή του συστήματος αυτού ηλεκτρονικής κλήσης βελτιώνει τις πιθανότητες που έχουμε να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Εάν οι χρήστες ε, χρησιμοποιούν ιδιωτικά συστήματα ή ταξιδεύουν σε χώρες όπου δεν υπάρχει αυτό το σύστημα, τότε θα πρέπει οι υπάροχοι, οι φορείς ε, τηλεπικοινωνιακοί να προσφέρουν αυτό αυτή τη δυνατότητα ούτως ή άλλως. Άλλωστε είναι πολύ σημαντικό και για την ενθάρρυνση της ε, καινοτομία στην Ευρώπη. Το έγνος, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση, ο Γαλιλαίος, ο Ευρωπαϊκός Διορυφόρος ε, αξιοποιούνται και μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις ευκαιρίες που μας δίδονται για να εφαρμόσουμε καλύτερα ε, το σύστημα αυτό. Ευχαριστώ. So, uh, now we can Ευχαριστούμε. Ολοκληρώνεται η διαδικασία Catch Να δώσουμε το λόγο τώρα στον ε, Επίτροπο κύριο Κάλλας για να ολοκληρώσει τη συζήτηση εκφράζοντας την άποψη της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικότερα τις Επιτροπές ε, Τραν Ίμκο και τους εισηγητές, ε, την κυρία Σενιάλοβα και τον κύριο Κόχ, για την δουλειά τους που οδηγήσει στην εξαιρετική αυτή έκθεση για το ECOL. Το ECOL είναι μία από τις ε, ε, δράσεις προτεραιότητας ε, στην οδηγία για τα συστήματα μεταφορών και θα συμβάλλει πάρα πολύ στην αύξηση της ταχύτητας και αποτελεσματικότητας της διάσωσης. Η εισαγωγή υπηρεσία υπηρεσίας ECOL με βάση των 112 είναι μια υψηλή προτεραιότητα της Κομισιόν και τη δουλεύουμε εδώ και κάποια χρόνια. Ε, χαιρετίζω την θερμή ε, υποστήριξη του Κοινοβουλίου που θα μέσα από την έκθεση που θα ψηφιστεί αύριο. Οι ε, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας ε, θα ρυθμιστούν το Σεπτέμβριο. Υπάρχουν και άλλες ε, οδηγίες που θα συμβάλλουν στο να γίνει λειτουργική λύση το 2015. Ε, πρέπει να ληφθεί υπόψη και η νομοθεσία ε, που διέπει την έγκριση του τύπου. Αυτή τώρα σχεδιάζεται και θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τους επόμενους μήνες. Οι προδιαγραφές για την αναβάθμιση των κέντρων απόκρισης ε, σε αυτές τις έκτακτες κλήσεις θα ρυθμιστούν στα πλαίσια της ε, ε, οδηγίας IPS. Σχεδόν έχουν οριστικοποιηθεί με τη βοήθεια ειδικών εμπειρογνωμόνων από όλη την Ευρώπη και η Κομισιόν θα οργανώσει αύριο την τελευταία συνάντηση των εμπειρογνωμόνων. Η έκθεση ζητεί υποχρεωτική εφαρμογή και ε, ανοίγει το δρόμο για την εναρμονισμένη χρήση των ε, ε, κλήσεων e-call με το 112. Ε, αυτό θα ισχύσει για όλους τους ενδιαφερομένους. Πιστεύω ότι η εφαρμογή υποχρεωτικά του e-call θα, επιτρέ... θα βοηθήσει να υπάρξουν οικονομίες κλίμακος και θα υπάρχουν ωφέλη όχι μόνο σε όλους τους πολίτες της Ευρώπης αλλά και στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Εμείς θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι τα απαραίτητα στοιχεία του e-call θα είναι λειτουργικά όταν θα εφαρμοστεί η υποχρεωτική χρήση του e-call. Όπως προτείνει η έκθεση, η Κομισιόν θα υποστηρίξει και την ενημέρωση ε, και την ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικές εκστρατείες, ούτως ώστε το e-call να χρησιμοποιείται σωστά. Θα προωθήσω την πλατφόρμα e-call και θα φροντίσουμε η επιλογή των πελατών και ο δίκαιος ανταγωνισμός να διασφαλίζονται. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνεχιζόμενη υποστήριξη στην χρησιμοποίηση και ανάπτυξη του e ώστε να γίνουν ασφαλέστεροι οι δρόμοι μας. Μαζί θα φέρουμε στους πολίτες του e για να σώσουμε πολύτιμες ζωές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Κλείνουμε τη συζήτηση αυτή και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις ε, 12 και 30. Προχωρούμε τώρα σε ένα άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη, ε, την έκθεση της κυρίας Ρόδης Κράτσα Τσαγκαροπούλου, ικανότητα προσέλκυσης επενδύσεων στην Ευρώπη. Και καταρχήν θα δώσω το λόγο